Äh, vielen Dank, äh, Kollegen. Workshop θα αρχίσουμε το workshop σχετικά με την ε, πολιτική σε σχέση με την γεωστρατηγική και το μέλλον της Αλφα και βεβαίως ξέρουμε ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες μέλη. Ο στόχος είναι ε, να σκεφτούμε μαζί και να εκπονήσουμε μια κοινή στρατηγική και πώς θα μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε ως εφαλτήρια τις εγκαταστάσεις τις οποίες έχουμε. Παραδείγματος χάρη ε, στο Τσάντα ε, και χωρίς ε, την ε, βάση που είχαμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στο τσάτο. ίδιο θα ισχύει και για την Σομαλία. Και βεβαίως μπορέσαμε να δράσουμε στο Τζιμπουτί. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να εκπροσωπηθεί στην Νότια Αφρική, στην Νότια Αφρική, στη Βόρεια Αφρική, ε, στην Οκεανία, ε, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι βάσεις που υπάρχουν και, με σημεία, και ως τα σημεία κίνησης και σαν εφαρτήρια αυτές οι βάσεις αποκτούν όλο και περισσότερο μεγάλη σημασία. Και βεβαίως η λευκή βίβλος αναφέρεται ε, στο Acte de Crise. Μπορούμε αυτή τη στιγμή με βάση το, την Ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλο να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, ποιες περιοχές υφίστανται μια κρίση ε, ποιοι κίνδυνοι ενέχονται και ποιες είναι οι δυνατότητες μας, ποιο είναι το δυναμικό μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να προβά, προλάβουμε στα μέτρα του δυνατού αυτές τις κρίσεις. Ε, έχουμε ανάμεσά μας τον δόκτωρα Σβέν Μπισκόπ, ο οποίος είναι διευθυντής του προγράμματος ασφάλισης και παγκόσμιας διακυβέρνησης στο Egmont Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων είναι αυτός ο οποίος θα κάνει μια εισαγωγή και επίσης έχουμε ε, ε, τον James Rogers, ο οποίος είναι υπότροφος επιστημονικής έρευνας στο Pembroke College του Cambridge και τον Λουίς ε, Σιμόνο, ο οποίος είναι υπότροφος του Thomas Holloway και συνεργάτης του προγράμματος σπουδών Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Και βεβαίως θα ε, αναφερθεί στον δυναμικό ρόλο που μπορεί να έχει η ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική και βεβαίως θα αρχίσουμε με τον δόκτορα Σβέν Μπίσκοπ, ο οποίος και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να απευθύνω το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πόσο μάλλον που απευθύνομαι σε πολύ διακυκρεμένους και ξεχωριστούς συναδέλφους. Νομίζω ότι ε, όσοι είναι διδακτορικοί υποψήφοι ή και κάτοχοι διδακτορικών ε, ήδη ζηλεύουν ε, εσάς για το βάθος των γνώσεών σας και της ανάλυσης που κάνετε εδώ. Σίγουρα το θέμα είναι κάπως αμφιλεγόμενο και σίγουρα υπάρχουν διάφορα ερετηματικά γύρω από αυτό μιλούμε για στρατιωτικές βάσεις και στρατιωτική παρουσία. Θα μιλήσουμε άραγε για τη διπλωματία των ε, πολεμικών ε, ελικοπτέρων ή σκαφών. Υπάρχουν αυτά τα ερωτηματικά. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να, να παραγνωρίσουμε την κατάσταση. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να έχει ένα εργαλείο και το σημαντικό είναι να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο θα το χρησιμοποιούμε καλύτερα. Το θέμα της ε, μελέτης αυτής εντάσσεται λοιπόν στην ευρύτερη ε, διαλογική σχέση που θα πρέπει να έχουν οι Ευρωπαίοι για το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσες είναι πραγματικά οι φιλοδοξίες μας. Έχουμε στρατηγική ε, για την ασφάλεια, έχουμε ένα κατευθυντήριο και βασικό στόχο. Έχω την εντύπωση όμως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλουμε και αυτό είναι πρόβλημα και για τη δική μας πολιτική ασφάλειας και άμυνας και είναι πρόβλημα και για το ΝΑΤΟ, διότι αν δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλουμε τότε ε, δεν μπορούμε να ε, το επιτύχουμε κι Μπορεί να ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό, σε ποια κλίμακα, πόσο πολύ θέλουμε να ε, αναλάβουμε αυτά τα ε, καθήκοντα. Ποια είναι λοιπόν τα καθήκοντα που θέλουμε να αναλάβουμε. Είναι οι στόχοι της Πετρούπολης, υπάρχουν στη συνθήκη του Άμστερνταμ και ευρύτερο ορισμός θα υπάρξει και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν τον αποκαλώ διευρυμένο ορισμό, Πιστεύω ότι είναι πιο λεπτομερής ορισμός συγκριτικά με το προηγούμενο περιεχόμενο του κειμένου. Ε, νομίζω ότι όλα συμπεριλαμβάνονται εκεί εκτός από τη συλλογική άμυνα. Οι ερμηνείες όμως ποικίλουν. Έχουμε τη διακήρυξη ε, και τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2008 Εκεί φαίνεται τι είναι αυτά τα οποία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να κάνει βράχη πρόθεσμα. Αναφέρεται η δήλωση αυτή σε όλα τα σενάρια πάνω στα οποία δουλεύουν οι στρατιωτικές ε, δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από αυτό το οποίο αποκαλούμε high intensity operations, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ορισμένα κρατημέλη θεωρούν ότι ε, μιλούμε για οπισθοχώρηση ως προς τις φιλοδοξίες μας. Άλλα κρατημέλη θεωρούν ότι έτσι οι φιλοδοξίες μας εκτείνονται πολύ περισσότερο. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν γνωρίζουμε ποιες ακριβώς είναι οι φιλοδοξίες μας. Εγώ νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε όλο το φάσμα της στρατηγικής ασφάλειας και άμυνας όπου δει, όπου αυτό είναι απαραίτητο, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο. Η στρατηγική ασφάλειας λέει ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη. Ένας πολύ φιλόδοξος στόχος είναι αυτός, χωρίς όμως να μπαίνει σε λεπτομέρειες η στρατηγική αυτή. Προτεραιότητα για τη δική μας πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει να είναι η δική μας γειτονιά, θεωρώ. Επομένως, ε, η δέσμευσή μας θα πρέπει να ισχύει ε, σε περιπτώσεις κρίσης, αλλά και μετά. Έχουμε το Λίβανο, έχουμε τη Γεωργία. Πώς θα το ερμηνεύσουμε όμως αυτό. Η γειτονιά θα περιλάβουμε και τις χώρες του κόλπου. Θα θεωρήσουμε ότι η γειτονιά μας είναι και η Κεντρική Ασία. Η υποσαχάρια Αφρική από την άλλη φαίνεται να είναι προτεραιότητα. Έχουμε τρεις ε, αυτόνομες ε, δράσεις εκεί που εκτιλήσονται. Είναι όμως αυτό αποτέλεσμα στρατηγικής επιλογής ή είναι αποτέλεσμα καλών ε, παλαιών δεσμών φιλίας και ειδικά βελγικών δεσμών φιλίας. Εν πάση περιπτώσει η υποσαχάρια Αφρική πρέπει να παραμείνει στόχος κατά την άποψή μου, γιατί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή, Άλλωστε, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αποκτήσει δύναμη και εξουσία να σταθεί στα πόδια της η Ένωση Αφρικανικών Κρατών. Τέλος, έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τις σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Και ε, ασχολούμαστε και με αυτό στη μελέτη μας. Έχουμε δράσεις στις ακτές της Σομαλίας κατά της πειρατείας για να προστατεύσουμε τις θαλάσσιες ε, ε, οδούς του εμπορίου. Από εκεί και πέρα, εάν πιστεύουμε στο σύστημα συλλογική ασφάλεια των Ηνωμένων θα πρέπει να αναλάβουμε το μερίδιο του βάρου που μα αναλογεί. Εάν συμβάλλουμε τώρα βέβαια σε κάθε αποστολή και δράση των Ηνωμένων τότε θα πρέπει να αναλάβουμε κατελάχιστον ορισμένα καθήκοντα και ορισμένε ευθύνες και αρμοδιότητε, Δηλαδή, να προστατεύσουμε και να μπορέσουμε να ε, καλύψουμε σε περίπτωση συγκεκριμένων πολλών και διαφορετικών σεναρίων χάρη σε ισχυρή ευρωπαϊκή πίεση, ε, διπλωματική πίεση υιοθετήθηκε η, αντίστοιχη, η αντίστοιχη αρχή σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Συν της άλλης, ε, τίθεται το ερώτημα σε ποια κλίμακα, πόσο, σε πόσο βάθος θέλουμε να φτάσουμε. Έχουμε το headline goal, το βασικό στόχο των 60.000, αλλά στην πράξη μιλούμε για ομάδες ε, παρέμβασης, battle groups, τις οποίες μετά δεν αναπτύσσουμε. Αλλά φαίνεται ότι ε, δεν είναι αρκετές οι προσπάθειές μας. Αν, μιλούσαμε, μιλήσουμε για όλες τις αποστολές ε, και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΝΑΤΟ ή Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κινητοποιήσουμε στρατεύματα 80.000, δηλαδή κάτι το οποίο ξεπερνά ε, ε, τον στόχο των 60.000. Άλλωστε, Έχουμε 1,8 εκατομμύρια ενστόλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι χρήσιμη όλη αυτή η ένστολοι στρατιωτική και μη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Το έγγραφο αυτό, κατά την άποψή μου, ουσιαστικά αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των ευρύτερων πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας ε, και της πρακτικής υλοποίησης και εφαρμογής. Θα μπορούσατε να θεωρήσετε ότι είναι μια λευκή βίβλος ή μια βασική στρατηγική ε, για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Είναι το έγγραφο που θα πρέπει να μας καθοδηγεί στις προσπάθειές μας, γιατί δείχνει πώς θα μετουσιώσουμε τους στόχους μας σε πράξη. Βέβαια το έγγραφο έχει τελείως ουδέτερη στάση ως προς την αιώνια αυτή ε, συζήτηση και διαλεκτική μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ε, πώς θα επιλέξουμε να δράσουμε ε, διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμέσου της πολιτικής της, ε, διαμέσου του ΝΑΤΟ ή διαμέσου των Ηνωμένων Εθνών, είναι έτερον εκάτερον. Θα πρέπει να επιλέγουμε κάθε φορά αναλόγως με το θέμα την περίπτωση. Σε άλλες περιπτώσεις αρμόζει καλύτερα να δράσουμε σε επίπεδο ΝΑΤΟ, σε άλλες αρμόζει καλύτερα να εφαρμόσουμε τη δική μας πολιτική γιατί το ΝΑΤΟ θα είναι αντιπαραγωγικό στην εκάστοτε περίπτωση. Το ΝΑΤΟ, ας πούμε, θα ήταν αντιπαραγωγικό στην ε, περίπτωση του Λιβάνου. Καλό είναι λοιπόν να μην δράσουμε μέσα από αυτό το διάβλο. Ως Ευρωπαίοι θα επιλέγουμε λοιπόν κάθε φορά και καλό θα ήταν πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, να αποφασίσουμε πόσο φιλόδοξοι θέλουμε να είμαστε πόσο φιλόδοξη θέλει να είναι αυτή η πολιτική. Άλλωστε, οι άλλοι εταίροι μας, οι Ηνωμένε Πολιτείε μεταξύ άλλων, περιμένουν από εμά να δράσουμε ε, ενιαία, να δράσουμε ενωμένοι. Τίθεται το ερώτημα γιατί θέλετε να προσδιορίσετε το επίπεδο στρατιωτικών φιλοδοξιών σας αφού αυτό έχει ήδη γίνει στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Νομίζω λοιπόν ότι η μελέτη αυτή δίνει απαντήσεις και έρχεται σε μια πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή από τη στιγμή που θα ξεκινήσει και θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση για το πόσο σημαντικός ε, παράγοντας θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα, στο στρατιωτικό σκέλος, στα στρατιωτικά θέματα. Θα πρέπει η Ευρώπη να προσέξει να μην χάσει την μπάλα, αντίθετα να κατορθώσει, να παίξει σωστά και να συμβάλλει σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος James Rogers. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή, την Υποεπιτροπή για την πρόσκληση που μας απίφθινε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Σβέν Μπίσκοπ διότι έκανε μια εξαιρετική σύνοψη και περίληψη της δουλειάς μας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα λεγόμενά του, διότι ταιριάζουν πολύ καλά με την εισαγωγική μου παρατήρηση. Στο παρελθόν οι εμπειρίες μας ήταν πολύ αρνητικές και γι' αυτό δεν ε, κατορθώσαμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη γεωστρατηγική. Ό,τι ελέγεται στην περίοδο του ψυχρού πολέμου είναι πλέον εκτός εποχής. Η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας και να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους μας σε έναν κόσμο πολλών και διαφορετικών πόλων. Άλλωστε το νέο περιβάλλον ασφαλείας επηρεάζεται από τους πολλούς και διαφορετικούς πόλους και κάτι το οποίο επηρεάζεται και από την δική μας στρατηγική. Ο επόμενος ομιλητής. Είναι σωστό, ε, μπορεί κανείς να πει ότι το 2003 έγινε η ανάλυση της στρατηγικής στα τέλη του 2008 όμως δημοσιεύτηκε η αξιολόγηση και σε αυτή την αξιολόγηση τονίζονται οι αλλαγές που έχει υποστεί το στρατηγικό μας περιβάλλον τα τελευταία πέντε χρόνια από την δημοσίευση της πρώτης έκθεσης το 2003. Μιλούμε λοιπόν για την ανάδυση κυρίως της Ασίας και για την επίταση της παγκοσμιοποίησης. Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν ιδιαίτερως και την εμπορική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την πολιτική της για την ασφάλεια. Η Ευρασία, όλη αυτή η ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται από τη διόρυγα του Σουέζ μέχρι και την Σαγκάη στον Ειρηνικό ωκεανό θα αποκτήσει όλο και περισσότερη σημασία ε, για την κοινή ευρωπαϊκή ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας τις επόμενες δεκαετίες. Θα ήθελα, λέει ο κύριος Ρότζες τώρα, να σας παρουσιάσω την ε, δομή της παρουσίασής μας, της εισήγησής μας. Έξι μέρη είναι αυτά που αποτελούν την ε, παρουσίασή μας. Θα συζητήσουμε για το ρόλο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων καταρχάς σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα μιλήσουμε για την ξένη παρουσία, για την απώλεια ισχύω, για τις ιστορικές διαστάσεις του θέματος. Άλλωστε, εμείς ήμασταν οι πρώτοι στην Ευρώπη που είχαμε ξένη παρουσία παγκοσμίω. Η Ευρώπη ήταν η πρώτη που είχε ξένη παρουσία ε, σε άλλες περιοχές στον κόσμο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου κυρίως και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τις στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις ή βάσεις και το ρόλο που θα διαδραματίσουν αυτές τα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια θα δούμε πώς ταιριάζουν όλα αυτά με τις ασύμετρες απειλές ασφάλειας. Ε, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, λαθρομετανάστευση και το καθεξής. Και τέλος θα προσφέρουμε κάποιες συστάσεις ε, χάραξης πολιτικής με βάση την ε, εισηγήσή μας. Ο κύριος Σιμών. Θα θέλαμε Καταρχάς να πούμε ότι η ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι παράδειγμα της γεωπολιτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές χρονικές περίοδοι. Ε, τρεις είναι οι βασικές εποχές που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή ε, γεωπολιτική διαδρομή. Η πρώτη είναι η εποχή από το 1952 με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα μέχρι και το 1992. Είναι η περίοδος της υπηρετικής ολοκλήρωσης, της ολοκλήρωσης της υπήρου, αν θέλετε. Και είναι η περίοδος συγκρότησης και δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας άνθησης εμπορικών δασμών στο διατλαντικό πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δεύτερη εποχή είναι η εποχή που εκτείνεται από το 1993, δηλαδή από την επικύρωση της συνθήκης του Μάστριτ μέχρι και το 2007. Και το επίκεντρο ε, τώρα πλέον είναι η παγίωση της οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στο επίκεντρο βρίσκεται η επέκταση των συνθηκών ασφάλειας και ευημερία της Ευρώπης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο με την προσχώρηση των ανατολικών χωρών. Άλλωστε έχουμε καταρχάς την προσχώρηση του 95 των πρώτων χωρών και των υπολείπων του 2004. Έχουμε τη διαδικασία της ε, Βαρκελόνης. Και σήμερα εξελίσσονται περαιτέρω οι πρωτοβουλίες αυτές με την εταιρική σχέση προς Ανατολάς και την Ένωση για την Μεσόγειο. Τέλος, θεωρούμε ότι η τελευταία εποχή της γεωπολιτικής διαδρομής στην Ευρώπη είναι αυτή που ξεκινάει από το 2007 και εκτείνεται μέχρι και σήμερα και ουσιαστικά είναι η παγκόσμια εποχή πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναδύονται ιδέες καινούργιε για την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, η οποία καταρχάς είχε γίνει αντιληπτή ως ένα πιο περιφερειακό πλαίσιο. Η παγκόσμια λοιπόν περίοδος, η παγκόσμια εποχή χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό πολιτικών και στρατιωτικών μέσων αλλά και διπλωματικών ώστε να επιτευχθούν καλύτερα οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Μιλούμε για μια νέα γεωπολιτική εποχή η οποία μας ε, κάνει να σκεφτόμαστε να μας κάνει να σκεφτόμαστε την έννοια της ε, παρουσίας μας στο εξωτερικό, αυτό το οποίο ονομάζουμε foreign presence. Είναι μια έννοια αυτή η παρουσία στο εξωτερικό, η οποία δεν ε, περιορίζεται στα στενά όρια της ύπαρξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε, ε, στο εξωτερικό. Αντίθετα, η παρουσία στο εξωτερικό είναι μια πολύ πιο ευρία έννοια με πολλές συνιστώσεις και προσωρινές και μόνιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό που μπορούν να στηρίξουν ε, δυνάμεις που θα αναπτύσσονται. Περιλαμβάνει επίσης δυνάμεις επίθεσης οι οποίες ε, έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό και μπορούν πολύ γρήγορα να κινητοποιηθούν και στο εξωτερικό. Περιλαμβάνει ε, δυνατότητες επιμελητίας, αφοδιασμού και υποστήριξης όλων των υπολείπων. Περιλαμβάνει δυνάμεις γρήγορης ανοικοδόμησης, οι οποίες μπορούν πολύ εύκολα να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο ε, συλλογικών εντολών Global Command, ε, συλλογικής και παγκόσμιας διοίκησης, γενικής διοίκησης όλων αυτών των υπόδομων και ένα βασικό δίκτυο ε, για την κεντρική επικοινωνία μεταξύ όλων αυτών των πτυχών, των ε, σκελών της ε, στρατιωτικής παρουσίας. Η εξωτερική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ε, είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Στην έκθεση του 2003 μιλούμε για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, για την ε, πάυση της χρήσης των όπλων μαζικής καταστροφής ε, και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχουμε ε, τις έννοιες της προληπτικής άμυνας, της συνολικής ασφάλειας και της σωστής ισορροπίας μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών εργαλείων, λέει ο κύριος Σιμών. Ο κύριος Ρότζες τώρα. Όλη, όλη αυτή η έννοια λοιπόν, η έννοια της παρουσίας στο εξωτερικό προέκυψε από τον Μπόλντεν το 1962, ο οποίος δεν ανακάλυψε την πυρίτιδα. Υπήρχε ήδη αυτή η έννοια και μπορείτε να δείτε τις απαρχές της στη μελέτη που σας έχουμε υποβάλει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί μπορείτε να βρείτε τα, όλα αυτά τα θέματα και τις λεπτομέρειες στο κείμενο, είναι άλλωστε πολύ περίπλοκο. Θα προσπαθήσω όμως να σας δείξω ε, πώς λειτουργεί αυτή η έννοια. Ας πούμε ότι έχουμε μια χώρα, την Blue Land, μια υποθετική χώρα, η οποία για να επηρεάσει ε, μια περιοχή στη Νότια Αμερική μπορεί να το κάνει. Όμως, εν τω μεταξύ, παρεμβαίνονται και άλλες χώρες. Έχουμε την Pinkland, για παράδειγμα, η οποία είναι στην σημερινή Βραζιλία, ενώ η Blue Land είναι στη σημερινή Γρυλανδία. Μπορεί κανείς να έχει λοιπόν διπλωματικές πρεσβείες ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βάσεις στην γειτονιά, σε μια φιλική γειτνιάζουσα χώρα, σε μια πρώην απικία ενδεχομένω. Μετά, έχει πρόβλημα εφοδιασμού η Blue Land. Πώς θα φτάσει τις μονάδες της να τις τροφοδοτήσει. Μπορεί να κατατρέχεται από το πολιτικό σύστημα στην Πίνκλαντ, στην ενδιάμεση χώρα. Και έχουμε έναν κύκλο επιρροών που δημιουργείται από την διπλωματική πρεσβεία. Βλέπετε το βέλος στην οθόνη και βλέπετε ότι με το βέλος σας δείχνω το σημείο στο οποίο η αλυσίδα εφοδιασμού και επιμελητίας πάσχει τον αδύναμο κρίκο. Πρέπει να περάσει από άλλες πρεσβείες ή από άλλες στρατιωτικές βάσεις για να φτάσει ε, η προμήθεια στην ενδιαφερόμενη μονάδα. Κάτι το οποίο καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά περίπλοκη. Άρα μιλούμε για μια πολύ μεγαλύτερη ε, σφαίρα επιρροής και τελικά η Blue Land μπορεί πιο εύκολα να επηρεάσει την, ε, να εξαρτάται ιδιαίτερως από την Land με τρόπους που πραγματικά ε, δεν της αρέσουν. Δηλαδή ακριβώς διότι πρέπει να περάσει μέσα από πολλά και διαφορετικά στοιχεία και σημεία της δεύτερης χώρας, γι' αυτό τον λόγο ε, δημιουργείται πρόβλημα. Σκεφτείτε το παράδειγμα της Πορτογαλίας η οποία είχε επεκτείνει τη σφαίρα της επιρροής της σε πολλούς και διαφορετικούς ωκεανούς ε, την εποχή εκείνη. Τότε μιλούσαμε για μια Ιβυρική Ένωση ουσιαστικά. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο σύστημα κυριαρχίας στην Βόρεια και Νότια Αμερική, αλλά και στην Αφρική, στην Ινδονησία, στην Ανατολική Ασία. Είχαμε όλες αυτές τις ε, διασυνδέσεις. Στη συνέχεια, τη θέση ε, της Ιβηρικής ε, επικράτειας κατέλαβε η Βρετανική Αυτοκρατορία και βλέπετε στην οθόνη τις γραμμές του τηλεγράφου, τους διάβλους επικοινωνίας, προμήθειας, εφοδιασμού. Βλέπετε στο χάρτη την έκταση της Βρετανικής Υπηρωής ανά τον κόσμο και είχαν φτιαχτεί τότε και ναυτικές βάσεις για να στηριχθεί το σύστημα αυτό και για να μπει σε μια τάξη, παρόλο που συχνά ήταν σε βάρος των γηγενών. Μιλούμε λοιπόν για την έννοια της απώλειας του, της βαθμίδας ισχύω. Αυτό είναι αυτό το οποίο ε, είχε ε, προβληθεί ως έννοια για πρώτη φορά το 1962. Τώρα, βλέπουμε κάτι που μας έχει δείξει πρώτα ένας Ολλανδοαμερικανός, ο Νίκολας Γκέιτσμαν ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ουσιαστικά έπρεπε σιγά σιγά να διηθήσουν και να μπορέσουν να επηρεάσουν ε, τις ε, προηγούμενες μεγάλες δυνάμεις την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βεβαίως όλα αυτά ε, θα γίνονταν με την αλληλεμπλοκή και δράση των μεγάλων δυνάμεων Γαλλία, Ρωσία, η Γερμανία μεταξύ άλλων. Και βλέπετε ότι όλοι πιέζουν και ασκούν πιέσεις για να έχουν πρόσβαση στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στους χώρους του κόλπου, στον, στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, αλλά και στην Ανατολική Ασία. Ο κύριος Σιμών. Προχωρούμε τώρα Ας περάσουμε τώρα σε μια ε, σύντομη επισκόπηση των ε, στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και που τις ε, χειρίζονται κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Το βασικό σύστημα υπάρχει στην υπηρετική χώρα, στη Γαλλία και αποτελείται από τρία υποσυστήματα προς νότων, και ανατολάς. Το πρώτο είναι προς δυσμάς, προς τον Ατλαντικό, προς τη Γουιάννα και τις Αντίλες όπου ε, είναι παρούσες οι ε, γαλλικές δυνάμεις. Προς Ανατολάς εκτείνεται προς την γαλλική πολυνησία στον Ειρηνικό. Ε, το δεύτερο σύστημα, η δεύτερη παρουσία, εκτείνεται μέχρι τη Σενεγάλη και την Γκαμπόν και με τον τρόπο αυτό φτάνει η γαλλική παρουσία μέχρι το δυτικό κομμάτι της Αφρικής. Και η τρίτη παρουσία βρίσκεται σε όλη τη Μεσόγειο, ε, συμπεριλαμβάνεται μέχρι και το Τζιμπουτί, ε, το οποίο ε, περιλαμβάνει το, το, μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών, Γάλλων στρατιωτών εκτός ε, ε, Γαλλίας ε, και συμμετείχε στις, στις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Κατόπιν υπάρχουν και καταστάσεις στο Αμπουντάμπι που διευκολύνουν τους Γάλλους στις επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή. Αυτή το εσωτερικό σύστημα πάει και προς τα κάτω, προς τη Ρεωνιόν και βλέπετε εδώ και μία διαφάνεια που δείχνει τις εγκαταστάσεις αυτές στην ίσο Ρεωνιών. Εξάλλου βαδίζει και κάτω ανατολικά προς τη Νέα Καλλιδονία, στον ε, νότιο Ειρηνικό. Και τώρα θα περάσουμε στη γαλλική παρουσία. Συμμεσχολείται στην αγγλική, στην βρετανική κατ' ουσίαν ε, που είναι παρεμφερής, ε, ξεκινάει στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτείνεται μέχρι τη Μεσόγειο, κυρίως μέχρι το Γιβραλτάρ Εκεί ε, δεν υπάρχουν πλέον μόνιμες δυνάμεις. Προχωράει προς τα κάτω και φτάνει μέχρι τα νησιά Φόλκλαντ, ε, τα οποία είναι η μεγαλύτερη κατάσταση Μεγάλης Βρετανίας, η υπερπόντια. Και αυτή είναι ε, μια προβολή από δορυφόρο, η οποία, μια εικόνα που έχει ληφθεί από δορυφόρο. Η δεύτερη από την Κύπρο μέχρι την Ερυθρά Θάλησα και κατ' ουσίαν εδώ μιλάμε για αμερικανικές ε, στρατιωτικές εγκαταστάσεις παρότι υπάρχει ε, και ε, μια μικρή βρετανική στρατιωτική παρουσία και φτάνει μέχρι την Νοτιοανατολική Ασία που έχει ως στόχο να στηρίζει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπερνάι για να στηρίξει και την κυβέρνηση. Όσον αφορά λοιπόν τι ε, στρατιωτικέ εγκαταστάσει των δύο μεγάλων, μεγαλύτερων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό από την Ισπανία που έχει και εγκαταστάσει ε, στι Κανάριε ε, νήσου, οι ευρωπαϊκέ δυνάμει έχουν και κάποιε μικρέ εγκαταστάσει στην Κεντρική Ασία που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Αυτέ όμω οι εγκαταστάσει δεν είναι μόνιμε, ενώ οι γαλλικέ και οι βρετανικέ στρατιωτικέ εγκαταστάσει υπάρχουν και πάρα πολλά χρόνια. Και αν θέλετε αυτό είναι και κάποια κατάλοιπα της ε, Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Θα ήθελα επίσης ε, να σας δείξω πώς το νέο γεωπολιτικό ε, περιβάλλον διαμορφώνεται και γίνεται όλο και πιο σαφές με την πάροδο των ετών. Βλέπετε στο χάρτη στην Ευρωπαϊκή, βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ιαπωνία αυτές ε, κατά τον προηγούμενο αιώνα ήταν οι πιο σημαντικές ε, δυνάμεις στον ε, αιώνα που βρισκόμαστε τώρα, ορισμένες εξ αυτών, κυρίως η Κίνα και η Ινδία, ε, θα είναι πολύ πιο δυνατές ε, από ό,τι ήταν κατά το παρελθόν. Είναι λοιπόν δυνατόν μετά από 20 ή 30 χρόνια, εξαρτάται βέβαια από οικονομικές προβλέψεις και άλλους ε, παράγοντες, οι δύο αυτές χώρες θα μπορούσαν να καταστούν οι σημαντικότερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου, να ξεπεράσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό κατά το 2025 περίπου που δεν είναι και τόσο μακριά. Μία εξ αυτών ε, θα μπορούσε να έχει ε, ε, μεγαλύτερη οικονομική απόδοση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ από κοινού. Θα ήθελα να σας δείξω, θα θυμάστε, μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ προσπάθησαν να κυριαρχούν σε την περιοχή από το Ηνωμένο μέχρι την Ιαπωνία. Και θα σας δείξω πώς το σύστημα αυτό λειτουργεί στην Ανατολική Ασία. Ένα σύστημα που κατά την άποψή μου θα είναι όλο και πιο σημαντικό για τις ΗΠΑ καθώς αυξάνουν όλο και μεγαλύτερη, ε, αποκτούν μεγαλύτερη εξουσία η Κίνα και η Ινδία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ε, διότι θα εμφανιστούν νέε δυνάμει σε τελείω διαφορετικά μέρη του κόσμου και όπω συνέβη και με τη Σοβιετική Ένωση κατά το παρελθόν και προς δυσμάσκεψη να το θα εμφανιστούν νέα συστήματα πολύ πιο σημαντικά. Έτσι λοιπόν το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών ε, επικεντρώνεται στην Ανατολική Ασία, ε, στην ναυτική βάση του Σαντιάγκο <clears throat> και αυτό θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει σε ένα σύστημα που πάει από την ακτή της, ε, σε όλη την ακτή της Ανατολικής Ασίας. Και αυτά, όπως ξέρετε, ε, αναγέρθηκαν κατά την εποχή του ψυχρού πολέμου ως ένας τρόπος για αναχέτηση του κομμουνισμού, όπως πίστευαν οι Αμερικανοί, έτσι ώστε να μην διεισδύσει αυτός ε, στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας. Η Ιαπωνία ιτήθηκε, είχε κατασκευαστεί αρκετές, αρκετούς εγκαταστάσεις, ε, ναυτικές εγκαταστάσεις. Και επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και τα νησιά, το Χαβάη, ε, το Pearl Harbor. Αυτές ε, είναι οι δύο σημαντικότερες βάσεις που στήριζαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ανατολική Ασία. Βλέπετε λοιπόν βλέπουμε το σύστημα, το σύστημα forward presence, πώς ακριβώς αυτό λειτουργεί. Βέβαια, αυτά ε, ε, έγιναν πιο περίπλοκα τελευταία χρόνια, γιατί επέτυχε μεγαλύτερη εξουσία η Κίνα, έχει επενδύσει στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάρτισαν ένα έγγραφο προς το Κογκρέσιο για να περιγράψουν πώς ακριβώς εξελίσσεται αυτή η εξέλιξη. Η Κίνα όμως έχει πρόβλημα, γιατί έχει τόσους πολλούς τέρους ε, εταίρους Ευρωπαίους ε, στην περιοχή και έχει μόνο μία ε, διέξοδο προς την θάλασσα που βλέπετε στη διαφάνεια. Αυτό βέβαια αποτελεί πρόβλημα γιατί όπως βλέπετε έχουμε εδώ τα στενά μαλάκα τα οποία είναι, έχουν, είναι πολύ στενά και πολύ βαθιά και σε κάποια σημεία όμως είναι πολύ ρηχά. Εάν τελικά περάσει από εκεί ε, κάποιο μεγάλο ε, δεξαμενόπλιο θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί κυρίως ε, πρόβλημα στην Κίνα γιατί όπως σας είπα θα μπορούσε πολύ εύκολα θα μπορούσαν τα στενά αυτά να μπλοκαριστούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση σύγκρουσης. Πρέπει κανείς λοιπόν κάπως να παρακάμψει τα στενά αυτά. Και βλέπετε ναυτικές βάσεις που φτάνουν μέχρι το Μπαγκλαντές και τη Βυρμανία και κάτω μέχρι τη Σρι Λάνκα, στις Εχέλες και καταλήγουν ε, στο λιμάνι Γκουάντα στο Πακιστάν, το οποίο το ανέγειρε η ε, κυβέρνηση της Κίνας και νομίζω ότι είναι ένας ε, από τους, ε, μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές βάσεις στην περιοχή. Αυτά έχουν στόχο να διευκολύνουν την ε, Κίνα στο να μπορεί να ασκεί περιοχή, εξουσία στην περιοχή γιατί αν κλείσει η ε, περιοχή εκεί, η θαλάσσια δίωδος, ε, τότε ε, θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα και για τους αγωγούς ε, στο μέλλον, έτσι ώστε να διεισδύσουν οι αγωγοί και μέχρι την Κίνα, το Πακιστάν, ε, τη Βυρμανία και τον Μπαγκλαντές. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η Ινδία ανησυχεί όλο και περισσότερο ε, για αυτό που θεωρεί ότι είναι περικύκλωση από την Κίνα. Και από ό,τι βλέπουμε η Κίνα έχει περικυκλώσει την Ινδία ε, ως σαλιγκάρι. Πολλοί Ινδοί ανησυχούν ότι η Κίνα προσπαθεί να τους εγκλωβίσει. Γι' αυτό λοιπόν η Ινδία προσπαθεί να ξεφύγει από αυτόν τον εγκλωβισμό ε, δημιουργώντας, δημιουργώντας ε, νέες ε, ναυτικές βάσεις στην Κοκοά που είναι πλέον η μεγαλύτερη στην Ινδία. Εκεί υπάρχει και εργοστάσιο αεροναυπηγικής. Προσπαθεί επίση να φτάσει και στην Κεντρική Ασία, συνεργαζόμενη μερικές φορέ με τη Ρωσία για να ανοίξει μια νέα αεροπορική βάση στο Τατζικιστάν. Εξάλλου έχει αναβαθμίσει ε, την παρουσία της στα νησιά Άντεμον. Ε, με τον τρόπο αυτό θα έχει μεγαλύτερο έλεγχο των στενών Μαλάκα. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό, γιατί υπάρχουν ε, πλέον όπως σας είπα, νέοι γεωπολιτικοί παράγοντες και στρατηγικές που κατά κάποιον τρόπο μοιάζουν ε, με τις παραδοσιακές δυνάμεις. Αυτά αρχίζουν να συσχετίζονται με τις ασύμετρες απειλές ε, που στην Ευρώπη έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία, κυρίως κατά τα τελευταία χρόνια. Και από αυτού θα σας μιλήσει ο συνάδελφός μου. Οι σχέσεις λοιπόν ανάμεσα στις ε, μεγάλες δυνάμεις ε, και τις ασύμετρες απειλές δεν είναι κάτι το καινούριο. Υπάρχει εδώ και αρκετούς αιώνες, ε, κυρίως κατά το 19ο αιώνα και κατά τον 18ο, ο συσχετισμός αυτός ε, ήταν προφανής. Ε, οι ασύμετρες όμως, ε, τα σύμμετρα φαινόμενα δεν αποτελούν μόνο απειλή, αποτελούν και ευκαιρία για τη συνεργασία των μεγάλων δυνάμεων. Μπορεί κανείς δηλαδή, να το ερμηνεύσει προς δύο κατευθύνσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιήσει την εξουσία της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ασύμετρες απειλές σε συνεργασία με όλες τις αναδυόμενες δυνάμεις. Η συνεργασία αυτή ανάμεσα στις ε, μεγάλες δυνάμεις μπορεί να καταλήξει σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη που έχουν τη δυνατότητα να αποκλιμακώσουν την ένταση ε, ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Και οι μεγαλύτερες ασύμετρες απειλές ασφαλείας ε, στην Ευρώπη είναι η τρομοκρατία, η πειρατεία, το οργανωμένο έγκλημα, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η λαθρομετανάστευση και αρκετές άλλες. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να εγγυάται την ασφάλεια ε, των θαλασσών που την περιβάλλουν. Και έτσι φτάνουμε στην ε, Μεσόγειο, ε, στον κόλπο και φτάνουμε και στις ε, πρώτες συστάσεις χάραξης πολιτικής. Είναι δηλαδή η ανάγκη να αντιμετωπιστούν ε, οι απειλές ε, προς τα ευρωπαϊκά συμφέροντα από τις ε, όμορες περιοχές, κυρίως όπως σας είπα στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μέση Ανατολή. Και τούτα μπορούν να γίνουν ενισχύοντας ε, τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Αφρική, στη Μαύρη Θάλασσα με χώρες όπως η Γεωργία, η Ουκρανία και η Τουρκία. Επίσης πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Μέση Ανατολή η προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ασφάλεια των ε, υδάτων αυτής ε, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ε, την σύσταση Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής έτσι ώστε τα ναυτικά κεφάλαια της Ευρώπης να απελευθερωθούν και πέρα από ε, τις όμορες χώρες. Προτείνουμε λοιπόν έναν ειδικό εκπρόσωπο για θέματα γεωστρατηγικής να οριστεί από τον είπα εκπρόσωπο της ΚΕΠΑ έτσι ώστε να προσφέρει καθοδήγηση ε, σε τέτοιου θέματα. Και ανάμεσα στις αρμοδιότητες αυτού του ειδικού εκπροσώπου ε, θα μπορούσε να είναι η λεπτομερής ε, παρουσίαση όλων των υπαρχών των ευρωπαϊκών κεφαλαίων με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή ε, βάσεις, σκάφη, στόλος και ούτω καθεξής. Και έτσι να υπάρξει μια δυνατότητα να ενσωματωθούν ενσωματωθεί όλο αυτό το δυναμικό κεφάλαιο ή δυναμικό αν θέλετε και να ολοκληρωθεί. Και το σύστημα αυτό, το δυναμικό αυτό, πρέπει να ε, συνδεθεί με το ε, επιτελείο εδώ στις ε, Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι όχι απαραίτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίω οι Ευρωπαίοι. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνει απαραίτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι κάτι μέσα στην Ένωση, κάτι που ε, πρέπει να απασχολεί του ακαδημαϊκού, του πολιτικού, και σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, οικουμενικό, που θα ε, βοηθήσει να είμαστε αποτελεσματικότεροι σε θέματα ασφαλείας και να επικαιροποιήσουμε λιγάκι και την έκθεση περί ασφαλείας που ε, δημοσιεύθηκε το Δεκέμβρη. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η περιοχή είναι η πιο επικίνδυνη, η πιο ευμετάβλητη. Αναφέρομαι στη ζώνη από το Σουέζ μέχρι τη Σανγκάη. Αυτή τη ζώνη που βλέπετε στη διαφάνεια περιλαμβάνει τη Μεσή Ανατολή, τμήματα της Κεντρικής Ασίας, τον Κάφκασο, την Ινδία, Νότιο-Ανατολική Ασία, και την Κίνα, ένα κομμάτι της Κίνας, όπου θα θυμάστε πριν από ε, δύο εβδομάδες είχαμε ένα επεισόδιο ε, ανάμεσα σε ένα κινέζικο και ε, ένα αμερικανικό σκάφος. Αυτή λοιπόν η περιοχή, όπως σας είπα, είναι επικίνδυνη για λόγους από πλευράς από τη σκοπιά της ισορροπίας μπορούν να εκραγούν πολλές συγκρούσεις ασύμετρες Εκεί θα παίξουν ρόλο οι μεγάλες δυνάμεις, η Κίνα, η Ρωσία, οι Ευρωπαίοι και οι Ηνωμένε Πολιτείες που έχουν, όπως είπαμε, συμφέροντα ε, και εγκαταστάσει ε, διάσπαρτες σε όλη την περιοχή. Βεβαίω ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, α μην ξεχνάμε, ότι η Ευρώπη πιο συγκεκριμένα έχει ένα τεράστιο δυναμικό που σας το παρουσιάσαμε και ίσως τελικά ε, καταλήξουμε σε ένα ε, ολοκληρωμένο σύστημα ε, να συνενωθούν, συνενωθεί το γαλλικό και το βρετανικό δυναμικό και θα είναι ισότιμο του αμερικανικού. Εξάλλου βλέπουμε ότι όλο αυτό το σύστημα φτάνει και μέχρι το νότιο ειρηνικό και στο νότιο Ατλαντικό, στην Αφρικανική ακτή Φτάνουμε μέχρι την Νότια Αμερική. Και έχουμε εγκαταστάσεις που είναι διάσπαρτες ε, σε αυτή τη ζώνη από το Σουέζ μέχρι τη Σονγκάη που σας περιέγραψα προηγουμένως. Το πιο σημαντικό είναι το Τιμπουτί και το Διέγκο Γκαρσία. που οι βάσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά και για πολιτικές. Γιατί αυτές οι περιοχές είναι εκείνες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα υποφέρουν από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου ε, υπάρχουν, εδώ τρέχουν και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Φτάνουμε μέχρι τον Μπουρνάι και την Ανατολική Ασία μέχρι τη Νέα Καλλιδονία στην Αυστραλία βορράς Αυστραλίας. Αυτό λοιπόν το σύστημα ε, προσφέρει κάποια γεωστρατηγική εικόνα που πρέπει να σκεφτούμε για τα επόμενα χρόνια. Ήδη υπάρχουν αρκετές ε, εγκαταστάσεις, αν αυτές λοιπόν κατά κάποιον τρόπο συσχετιστούν και μπουν κάτω από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως ε, θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις ESDP. Και έτσι πρέπει να σκεφτούμε και τα θέματα της επιμελητίας. Οι Ευρωπαίοι, όπως ε, και άλλες μεγάλες δυνάμεις, ή σε σχέση με άλλες μεγάλες δυνάμεις, ε, δεν έχουν ε, μεγάλη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, χρησιμοποιούν τα σκάφη. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε κατά τα επόμενα έτη. Να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το στόλο, να είναι αποτελεσματικός, να συσχετιστούν με μονομένη στόλοι, να ολοκληρωθούν για να υπάρχει δυνατότητα άσκησης πολιτικής επιρροή... σε μια περιοχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέροντα. Αναφέρομαι κυρίως ε, στην ε, όμορφη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάποια ε, κομμάτια της Αφρικής και όλο και περισσότερο σε αυτή την περιοχή η Σουέζ Σανγκάη που παρεπιπτόντως είναι η περιοχή εκείνη όπου έχουμε τις βασικές ναυτικές οδούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, ε, Μεσόγειος ε, και πάλι προς τη Βόρεια Ευρώπη, τα μεγάλα λιμάνια στις ακτές της Ολλανδίας, της Μεγάλης Βρετανίας, ε, της Γαλλίας, της Γερμανίας. Και έτσι τελειώσαμε με την παρουσίασή μας και ελπίζουμε να σας άρεσε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη. Ε, μας δίνει έναυσμα για περαιτέρω σκέψη. Καταρχήν, το θέμα του ιστορικού. Βεβαίως ε, βρήκαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την ιστορική επισκόπηση και μόνιμο στοιχείο είναι βέβαια ότι δεν ισχύει μόνιμα ένα σύστημα. Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ότι σε αυτή την ε, Επιτροπή θέλουμε να ορίσουμε ποια είναι τα ενδιαφέροντα, τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εκπονήσουμε την στρατηγική μας επί τη βάση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Και βεβαίως εδώ εντάσσονται θέματα που άπτονται της ε, ασφάλειας, ε, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την προμήθειά μας σε ενέργεια. Θα πρέπει όλα αυτά να τα μελετήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε όλους αυτούς τους τομείς. Αν αυτό θα το κάνουμε σε συνεργασία με άλλους εταίρους, πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις που έχουμε και ε, βεβαίως θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι το δυναμικό ε, που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ο James Rogers αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, αναφέρθηκε δηλαδή στο δυναμικό, στις ικανότητες που έχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένες χώρες, αλλά όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα της στρατηγικής θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, πού θα δώσουμε το βάρος. Και βεβαίως υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, υπάρχουν Γάλλοι και Άγγλοι συνάδελφοι οι οποίοι ε, επιμένουν ε, Europe is a global power, η Ευρώπη αποτελεί μια δύναμη συνολική ε, και βεβαίως global power μπορούν να είναι και οι 60.000 στρατιώτες ε, και βεβαίως ε, δεν ξέρω το global power μπορούμε να το μεταφράσουμε ε, και σε οικονομικούς όρους. Λοιπόν, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας, για την συμβολή σας. Πιστεύω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έναυσμα για την συζήτησή μας και βεβαίως και για την συζήτηση που θα διεξαχθεί στο μέλλον ε, σχετικά με τη λευκή βίβλο που αναφέρεται στο θέμα της ασφάλειας και της άμυνας. Θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ συγκεκριμένα με αυτά τα ζητήματα. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική βάση για τη συζήτησή μας. Ο Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε που τόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις διεξάγονται στο τέλος της θητείας μας μόνο. Ελπίζω όμως ότι τα μέλη του επόμενου Κοινοβουλίου, κατά την επόμενη θητεία, θα συνεχίσουν αυτό το έργο και θα στεγάσουν και άλλες τέτοιες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Το είπατε κι εσείς ε, κύριοι ομιλητές. Οι βάσεις αυτές και οι εγκαταστάσεις αυτές είναι κατεξοχήν γαλλικές και βρετανικές, επομένως αντικατοπτρίζουν κυρίως τα, συμφέροντα αυτών των χωρών. Το θέμα είναι πόσο ε, μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, πόσο θα έρθουν πιο κοντά σε εμάς τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ή πόσο μπορεί να χτίσει πάνω στα προϋπάρχοντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο. Έχετε δίκιο και πολύ σωστά το δείξατε. Ε, όταν είναι κανείς μέλος μιας ένωσης, ε, αποκτά και περισσότερες ευθύνες και οι ευθύνες πολλαπλασιάζονται με την προσχώρηση ε, και άλλων κρατών μελών. Βεβαίως με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θέλει δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράγοντας στην Μαύρη Θάλασσα. Και αυτό είναι σημαντικό διότι ε, πρέπει να ασχοληθούμε με το εξή θέμα. Τι είδου βάσει θα πρέπει να φτιάξουμε στο μέλλον για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών δυνάμεων ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Θα πρέπει να έχουμε μόνιμε βάσει ή εγκαταστάσει. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να λύσουμε τα διάφορα επιχειρησιακά και λειτουργικά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούμε, το modus operandi, το μείγμα, τη συνταγή μεταξύ στρατιωτική παρουσία και ε, παρουσία πολιτικών δυνάμεων, μη στρατιωτικών, εν πάση περιπτώσει. Ε, Πάντοτε κανείς όταν μπαίνει σε ένα παιχνίδι πρέπει να μπαίνει και να παίζει σύμφωνα με τους κανόνες και πριν φτιάξει ένα παιχνίδι θα πρέπει να θέσει τους κανόνες. Και δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει συνειδητοποιήσει αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Εάν μιλούμε για προσωρινές βάσεις, για μη μόνιμες βάσεις, τότε έχουμε το πρόβλημα της προβολής των εξουσιών και το πρόβλημα της στήριξης του εφοδιασμού και της επιμελητίας. Βεβαίως ε, μπορείτε εσείς να αναφερθείτε στο περιβόητο Airbus Α400 και το καθεξής, αλλά τίθεται το ερώτημα πόσο μπορούμε εμείς να στηρίξουμε αυτή την προβολή εξουσίας, δύναμης, ισχύω αν θέλετε εκ μέρους κάποιων. Τέλος, Σίγουρα θα έχουμε αποστολές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Αποστολή π.χ. για την προστασία των θαλάσσιων επικοινωνιακών διάβλων. Και είναι κάτι που ήδη κάνουμε και κυρίως στον Ειδικό ωκεανό με το πρόβλημα της πειρατείας μεταξύ άλλων. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και το πρόβλημα της προστασίας των κρισίμων υποδομών μας. Η μεταφορά ενέργειας για παράδειγμα πρέπει οι ενεργειακοί μας πόροι να κατοχυρώνονται, να προστατεύονται και με στρατιωτικές δυνάμεις. Και συν της άλλης θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά και την αντίδρασή μας στις ανθρωπιστικές κρίσεις. Ε, κάτι το οποίο είναι τελείως ξεχωριστό, τελείως διαφορετικό. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας να καταφέρει να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα βασανιστικά ερωτήματα. Σας Ευχαριστώ. Ε, εδώ υπάρχει κάτι το περίεργο από την Πορτογαλία. Λοιπόν, τι έχει μείνει από τα παλιά πορτογαλέζικα συστήματα που είχατε εκεί. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστώ θερμά. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ε, και να σας συγχαρώ, Κάρλ, γιατί εσείς, Κάρλ, ε, διοργανώσατε στην τελευταία μας συνεδρίαση μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία θα μας εμπλουτίσει με πολλές και διαφορετικές σκέψεις και σίγουρα τη σκητάλη θα πάρουν οι συνάδελφοι που θα μας διαδεχθούν μετά τις εκλογές. Δεν ήμουν παρούσα ε, προηγουμένως όταν έγινε αναφορά στη δουλειά που κάνατε εσείς, Καρλ, στη δουλειά της ε, Προεδρίας της δικής μας Επιτροπής. Ε, δράτω με λοιπόν τις ευκαιρίες να σας συγχαρώ για την Προεδρία σας. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να εργαστώ δίπλα σας Νιώθω ότι η υποεπιτροπή μας βιώνει την πολύ έντονη ανάγκη να εμπλουτίσει τις γνώσεις της, να μάθει πολλά περισσότερα για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική. Αυτά τα πέντε χρόνια πιστεύω ότι έχουμε επιτελέσει ένα σημαντικό έργο με τη δική σας βοήθεια προς όφελος της Ευρώπης. Και λυπούμε πολύ διότι τόσοι λίγοι συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατανοούν πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα θέματα στρατηγικής και τακτικής τα οποία συζητούμε εμείς εδώ στη δική μας Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Από εκεί και πέρα, ε, κατά την άποψή μου, το πεδίο στο οποίο εμβάθυνα τις γνώσεις μου ε, κατάφερα ακριβώς να κάνω αυτό, να πετύχω αυτό το αποτέλεσμα χάρη στην ύπαρξη αυτής της υποεπιτροπής. Διότι ε, συνειδητοποίησα ότι οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί που θα πρέπει να εμπλέκονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, θα πρέπει να τους δοθούν πολύ περισσότερες δυνατότητες. Εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να χαράσουμε τις εξελίξεις στα θέματα ασφαλείας και άμυνας, γιατί είμαστε αιρετοί και θα πρέπει λοιπόν να μας περιλαμβάνουν πολύ περισσότερο στις συζητήσεις τους οι διάφοροι ηθήνοντες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και εκτός Κοινοβουλίου στις διάφορες καθεστικίες τάξεις πολιτικές και στρατιωτικές ανά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ συχνά χανόμαστε σε αυτή την ανόητη διαμάχη κατά την άποψή μου. Ποιο πλαίσιο ταιριάζει καλύτερα για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρώπη, το πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό για μένα είναι να ξεπεράσουμε επιτέλους αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή έχει κλείσει τον κύκλο της τον έχει κάνει τον κύκλο της λοιπόν, τον έχει κλείσει και να προχωρήσουμε ε, περαιτέρω. Έγινε μια συνάντηση πρόσφατα ε, στις Βρυξέλλες ε, μεταξύ Βρετανών και Γερμανών αλλά και άλλων με βασικό αντικείμενο τι διγενέστε για να ενισχύσουμε το στρατιωτικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η προφανής απάντηση είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία δεν ε, αποτελεί, ούτε σχετίζεται, ούτε εξαρτάται μόνο από τον απλό στρατιωτικό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Πρέπει λοιπόν να ξεκολλήσουμε από αυτή τη συζήτηση και να προχωρήσουμε ε, παραπέρα. Άλλωστε και η δική μου πολιτική ομάδα, οι σοσιαλιστές, το παραδέχομαι. Ε, είχαμε εμπλακεί σε άλλες ατραπούς, αν θέλετε, στο παρελθόν. Ε, είχαμε κολλήσει με τις αντελήψεις μας και δεν είχαμε τη σωστή στάση για τα θέματα αυτά. Στο θέμα μας τώρα, στη συζήτηση τη σημερινή. Να πω καταρχάς ότι δεν συμφωνώ απαραίτητο με τον κατάλογο των απειλών και δεν συμφωνώ με τη συμπερίληψη της λαθρομετανάστευσης σε αυτό τον κατάλογο των ασύμετρων απειλών. Νομίζω ότι ε, εάν βάλουμε την λαθρομετανάστευση την ίδια ζυγαριά με το οργανωμένο έγκλημα ή την τρομοκρατία, ε, θα έχουμε πρόβλημα. Ξέρετε, η Ευρώπη είναι προϊόν της λαθρομετανάστευσης. Ε, είναι κάτι που χαρακτηρίζει Νομίζω ότι είναι πολύ μειωτικό να συμπεριλάβουμε τη λαθρομετανάστευση στις ασύμετρες παγκόσμιες απειλές για την ασφάλεια. Είναι απλούστευτικός τρόπος σκέψης. Είναι κάτι το εσφαλμένο, κατά την άποψή μου. Βεβαίως δεν εννοώ ότι εάν η λαθρομετανάστευση σχετίζεται με ποινικό κολάσιμε δραστηριότητε, αυτό δεν είναι απειλή. Βεβαίω και είναι απειλή. Αυτό το παραδέχομαι. Όμως το οργανωμένο έγκλημα είναι κάτι το πολύ πιο σοβαρό. Άλλωστε η μετανάστευση ανέκαθεν αποτελούσε ελαθρέα ή και νόμιμη ε, μια βασική ζωτική δύναμη για την ανακατανομή των εσχή, των δεξουσιών στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, όντως δεν έχουμε ναυτική στρατηγική η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία ασφαλείας. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Στρατηγική, στρατηγική για τη θάλασσα ευρύτερα, αλλά δεν έχουμε περιλάβει τα θέματα ασφαλείας. Και συμφωνώ με τον κύριο Πασκούντο, ο οποίος είπε ότι οι μηχανισμοί που διαθέτουμε βασικά είναι γαλλικές και βρετανικές βάσεις, οι οποίες καθόλου δεν σχετίζονται με την ευρωπαϊκή λογική, αντιθέτως σχετίζονται με την γαλλική και βρετανική λογική αντιστοίχως. Η σημερινή στρατηγική μας για τα ναυτικά θέματα δεν δίνει τη βάση που χρειάζεται ε, στα θέματα ασφαλείας. Αυτό είναι σίγουρο και συμφωνώ μαζί σας. Επίσης, δεν αναφερθήκατε και σε ένα άλλο στοιχείο, την κυβερνοπειρατεία, η οποία αποτελεί βασική ε, πράξη ε, διάρρηξης του κοινωνικού ιστού και πλήγματος των οικονομιών μας. διότι σχετίζονται όλα αυτά τα αγαθά και με την κυβερνοπειρατεία. Η κυβερνοπειρατεία μπορεί να πλήξει και τα ενεργειακά μας αγαθά, αλλά και άλλα. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσετε αυτό το θέμα, να μάθω τις απόψεις σας για την κυβερνοπειρατεία. Επιπλέον, η μελέτη σας βασίζεται στην εξής ε, κύρια παραδοχή, ότι η πρόσβαση στο πετρέλαιο είναι εξαιρετικά σημαντική, κάτι και για τη ΣΥΠΑ και για την Κίνα και για όλους. Όμως, η παραδοχή αυτή δεν σημαίνει ότι είναι και το ε, θέσφατο. Ίσως ε, είμαστε πρώτον πυλών και ίσως έρθει, δημιουργηθεί ένας καινούριος κόσμος όπου δεν θα εξαρτώμεθα τόσο πολύ από το πετρέλαιο, θα έχουμε πολύ πιο ε, πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα τις αξιοποιήσουμε καλύτερα. Επομένως η ανάγκη ε, η πετρελαϊκή θα είναι ε, πολύ λιγότερο σημαντική και πολύ περισσότερο σημαντικά θα είναι άλλα πράγματα όπως είναι ας πούμε, η διαδικτυακή ασφάλεια μεταξύ άλλων. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσετε αυτά τα θέματα. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για τη καλά σας λόγια, ο κύριος Τζέφρι Φον Χόγκιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ο λόγος για τον οποίο γίνεται λόγος για την ε, λαθομετανάστευση και εξισώνεται αυτή με την τρομοκρατία είναι ότι η ε, λαθρομετανάστευση είναι εκείνη που καθιστά ε, τροτή την ε, εθνική μας ταυτότητα. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διορτηθούμε από πού προέρχονται όλα αυτά. Δεν μπορούμε ε, τα δύο αυτά θέματα να τα διαχωρίσουμε. Εκείνο το οποίο περιγράψατε ως αστεία διαμάχη δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι θεμελιώδης. Και αυτή είναι και μία από τις παρατηρήσεις που θέλω να κάνω για τις ομιλίες που ακούσαμε. Δεν γίνεται καθόλου αναφορά στο ΝΑΤΟ. Και πρέπει να πω δεν ξέρω αν αυτή η ομιλία ήταν ε, ε, έτσι ε, σχεδιασμένη. Αν είχε λάβει χώρα την 1η Απριλίου θα την είχα καταλάβει. Θα ήταν μέσα στο σωστό πλαίσιο. Όμως ποτέ δεν έχω ακούσει τέτοιου είδους παρουσίαση των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολλές φορές ε, για αστείο ε, λέμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει τη σημαία της στους δικούς της τους στρατιώτες. Τώρα λέμε ότι θα πρέπει να βάλει τη σημαία της στις Βρετανικές και άλλες βάσεις ανά τον κόσμο. Αυτό πραγματικά το βρίσκω πολύ τραβηγμένο. Όσον αφορά τη δική μας την ασφάλεια, τη σκεφτόμαστε πάντα σε σχέση με το ΝΑΤΟ και τις δημοκρατίες. Γιατί οι δημοκρατίες είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν τις ε, προκλήσεις και οι δημοκρατίες ε, πρέπει να σκεφτούν πώς μπορούν να υπερκεράσουν αυτές τις ε, προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις. Ε, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει το δικό της το στίγμα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις που ήδη αναπτύσσονται σε κάποιο άλλο σημείο του κόσμου. Και δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι η ε, προστιθέμενη αξία αυτού που κάνετε. Από ό,τι βλέπω εγώ δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να σταματήσει τη Μεγάλη Βρετανία, τα κύματα. Ο κύριος Φόντιν, ο επόμενος ομιλητής. Θα ήθελα να εμφωνήσω ε, βεβαίως όλα αυτά που λέξαμε μέχρι τώρα για το δικό σας ε, το ρόλο. Εν πάση περιπτώσει ε, θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε. Και θέλω επίσης να πω ότι ο κύριος Βαν Όρντεν πήρε τη δόση του, της οργής. Ξέρουμε πολύ καλά από που προέρχεται. Εδώ δεν πρόκειται για ανάλυση του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται για μια ανάλυση του τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη ε, την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε βρετανικές βάσεις. Ο κ. Βαν Όρντεν μπορεί να μην το θυμάται, αλλά είμαστε όλοι ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εγώ ε, είχα την εντύπωση ότι το Γιβραλτάρ περισσότερο είναι επικράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι υπερπόντια περιοχή. Θα το δούμε την επόμενη φορά, θα τους το πω και ίσως μπορούμε από αυτό να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη. Πρέπει λοιπόν να πω ότι και εγώ έχω ε, κάνει κάποια δουλειά για τη βάση Diego Garcia. Είναι δύσκολο να πει κανείς ότι είναι Βρετανική βάση. Είναι Αμερικανική βάση με κάποιους ε, Βρετανούς που περιφέρονται. Οι Αμερικανοί έχουν βάλει τη δική τους την σημαία σε ε, Βρετανικό έδαφος. Φαντάζομαι ότι και αυτό θα εξοργίζει τα μάλα των κύριο Βανόρντεν. Και νομίζω ότι Ίσως αυτό ε, βοηθήσει και κάποια νησιά να επανέλθουν ε, στην ε, επικράτεια της Βρετανίας. Τέλο πάνω, δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό εδώ. Η δική μου βασική ερώτηση αφορά στις, στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ποιοι θα είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι το 2050. Αυτή είναι η ερώτησή μου συνάδελφος Λαντσμπέργκης. Και εγώ θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία για να μου διευκρινίσετε κάποιες έννοιες, για να καταλάβω κάτι. Και η επόμενη ερώτησή μου είναι η εξής. Μας παρουσιάσατε τις εξελίξεις στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύο φάσεις ολοκλήρωση και κατόπιν ε, επέκταση και παγίωση. Και οι δύο αυτές έννοιες έχουν πολιτικό βάρος και ουσία. Πώς πρέπει κανείς να ερμηνεύει αυτή την ε, υπηρετική ολοκλήρωση. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμα απόλυτα υπηρετική είναι κατά το ίμιση. Υπάρχουν και οι υπερπόντιες περιοχές ως έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Κατόπιν, η επόμενη φάση είναι η επέκταση και η παγίωση από το 1993 μέχρι το 2007 η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη κατά αυτήν την περίοδο. Ίσως λοιπόν δεν είναι καλή αυτή η διατύπωση περί επέκτασης. Εγώ δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επεκτατική δύναμη. Υπό την προπόθεση βέβαια ότι αυτό αποτελεί και συγκεκριμένη πολιτική. Γιατί λοιπόν δεν χρησιμοποιείτε τη λέξη διεύρυνση. Ίσως ε, γίνεται λόγος για την επέκταση σε υπερπόντια εδάφη. Τώρα μιλάμε περισσότερο για ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αν δει κανεί και τα Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής. Όμως, κατά την πρώτη περίοδο ε, δεν ε, είχαμε υπηρετική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Βεβαίως, αν χρησιμοποιείτε αυτή την έννοια ως ε, αντιπαραβολή στα υπερπόντια εδάφη, τότε δεν ξέρω αν έχετε αυτό κατά νου. Κατόπιν, δεν θα έλεγα για υπερπόντια παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως για παγκόσμια οικουμενική παρουσία με μεμονωμένων κρατών μελών ή της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς ε, ε, παρουσιάσατε πολύ ανάγλυφα όλη αυτή την κατάσταση και αναφερθήκατε και στην παρουσία των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ινδίας. Δεν αναφερθήκατε όμως στη Ρωσία. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην παρουσία της Ρωσίας. Η Ρωσία δεν έχει μόνο ε, ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις στη Μολδαβία, στη Γεωργία, στην Αρμενία έχουν και εγκαταστάσεις, ε, οι βάσεις στην Αρκτική, ε, ισχυρίζονται ακόμα και στο Βόρειο Πόλο και ε, προγραμματίζουν εγκαταστάσεις στη Βαλτική. Άρα δηλαδή υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας που θα υπάρξουν κατά το μέλλον και νομίζω μόνο έτσι έχει κανείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Και γι' αυτό ρωτώ γιατί αποφύγατε να θίξετε αυτό το θέμα των εγκαταστάσεων της Ρωσίας. Πρόεδρος, από ό,τι βλέπω δεν επιθυμεί κανείς άλλο το λόγο. Ε, θα θέλω λοιπόν να δώσω το λόγο στον πρώτο μιλητή. Ναι, δεν θέλω να καταλάβω όλο το χρονικό περιθώριο που μας έχετε δώσει. Γι' αυτό θα απαντήσω μόνο στο ερώτημα για τους συμμάχους. Αυτό σχετίζεται με την συζήτηση του πώς χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, αυτό το καινούριο εργαλείο, ενώ χτίζονται τέτοιου είδους σχέσεις παντού στον κόσμο ούτως ή άλλως. Έχουμε οικονομικές εταιρικές σχέσεις αλλά στα θέματα που μας ενδιαφέρουν ουσιαστικά δεν έχουμε εταιρική σχέση, έχουμε στρατηγικό διάλογο. Μιλούμε πολύ για αυτά, αλλά δεν κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, δεν πράττουμε πολύ μαζί. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να δώσουμε χώρο για αυτό το δεύτερο πυλώνα των εταιρικών σχέσεων που σας ανέφερα και προηγουμένως. Τίθεται το ερώτημα ποιος από αυτούς τους εταίρους είναι πιο φιλικός, διακείμενος προς ε, αυτό που θέλουμε εμείς να επιτύχουμε. Και πολλοί λένε ότι η απάντηση είναι ότι είναι οι Νοτιοαμερικάνοι. Η Βραζιλία, οι χώρες Λατινικής Αμερικής και το καθεξής. Είναι πιο εύκολο να σφυριλατήσουμε συμμαχίες με αυτούς. Άλλοι θα πούν ότι αυτός ο εταίρος είναι η Κίνα ή και η Ινδία. Μιλήσατε για τη συμμαχία των δημοκρατιών. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό γιατί πιστεύω ότι ε, το ρόλο αυτό τον επιτελούν τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ινδία είναι δημοκρατία, αλλά δεν λειτουργεί απαραίτητα με τον ευρωπαϊκό τρόπο. Έχει διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικό τρόπο σκέψης. Δεν νομίζω ότι η έννοια του forward presence, της παρουσίας στο προσκήνιο, αν θέλετε, στο εξωτερικό, ε, δεν περιλαμβάνει μόνο αυτό, περιλαμβάνει και τις εταιρικές σχέσεις με τους υπολείπους ε, εταίρους και παράγοντες στο παγκόσμιο ε, στερέωμα. Ο κύριος Σιμών τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως προς το πρώτο ερώτημα σας, ε, θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, είπατε ότι οι βάσεις είναι βασικά γαλλικές και βρετανικές και όντως έχετε δίκιο. Εμείς ήρθαμε για να κάνουμε μια στρατηγική επισκόπηση εδώ και γνωρίζουμε τα πολύ ουσιώδη πολιτικά εμπόδια σε αυτό που προτείνουμε. Ε, απλά θέλαμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή ακριβώς σε αυτό. Δεν μπορούν τα κράτη-μέλη από να τους να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους σε παγκόσμια κλίμακα, το καθένα μόνο του. Αυτό είναι σαφές είναι σαφές από την σύσταση των Ηνωμένων και την ίδρυση του ΝΑΤΟ. Και ανέκαθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να κρυφτεί πίσω από τη ΣΥΠΑ και να ε, επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην οικονομική και πολιτική της ανάπτυξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε προχωρούν προ τα ανατολικά για πολλού και διαφορετικού λόγου, μεταξύ των οποίων ο τελευταίο και πιο πρόσφατο λόγο είναι και η χρηματοπιστωτική κρίση. Υπαναχωρούν λοιπόν οι Ηνωμένε Πολιτείε και έχουμε εργαλείο, ε, είναι ένα εργαλείο αυτό, έχουμε μια ευκαιρία να καλύψουμε το κενό που θα αφήσουν. Γνωρίζουμε τα πολιτικά εμπόδια, αλλά μπορούν να υπερπηδηθούν κατά την άποψή μα. Ο κύριος Ρότζε τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το εξή: Μιλήσατε, μίλησε ένας ερωτών για το παιχνίδι για το αν οι Ευρωπαίοι πραγματικά θέλουν να παίξουν το γεωπολιτικό παιχνίδι, για το αν ξέρουν να παίζουν και θέλουν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, πώς αντιμετωπίζουμε την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν αντιμετωπίζουμε τους παίκτες αυτούς ισότιμα ή εάν ε, θα άλλη άποψη για τα πράγματα. Θα έλεγα λοιπόν ως απάντηση ότι δεν υπάρχει ίσως άλλη άποψη εάν κανείς δεν καταλαβαίνει πρώτα τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι παίκτες. Αν αυτό που θα κάνουν είναι κατά των προτεραιοτήτων σου ή των φιλοδοξιών σου ή των επιθυμιών σου ή οτιδήποτε, ε, τότε θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και να κοιτάξεις να, πέσεις το, να παίξεις το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, χωρίς όμως να θέσεις εν κινδύνο τις δικές σου επιδιώξεις. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε σε θέση να έχουμε την επισημία, να υπερασπιστούμε ε, τα επιχειρήματά μας και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί σε αυτή την καινούργια ισορροπία δυνάμεων, η οποία θα δημιουργηθεί ε, μέχρι το 2050, ε, όποτε και θα έχουν τελείως διαφορετικό ρόλο η Κίνα και η Ινδία. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε ε, την κατάσταση σήμερα. Είναι σαν να λέμε ότι μια μικρή αφρικανική χώρα θα αποκτήσει τη δυσχή των ΗΠΑ το 2050. Όμως γίνονται αυτές οι αλλαγές σιγά σιγά. Ε, η Κίνα θα αναδύεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο ως διεθνής παίκτης, η Ινδία το ίδιο. Ε, υπάρχει και η αλληλεμπλοκή με τη Ρωσία, η οποία θέλει να κατοχυρώνει όλο και πιο έντονα τη θέση της και την παρουσία της. Αυτό φαίνεται τα τελευταία δέκα χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν θα κλιμακωθούν κάποια στιγμή και θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ευρώπη χωρίς την Αμερική, ε, πρέπει να σας πω ότι νιώθω έτσι κάποια απογοήτευση ε, για το που βρίσκονται τα προβλήματα σε αυτή τη ζώνη από το Σουέζ μέχρι Σανγκάη. Υποτίθεται το Μεξικό και η Βραζιλία θα είναι τα προβλήματα. Ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Κάπου αλλού θα πρέπει να ψάξουμε να τα βρούμε. Εμείς βέβαια πρέπει να παίξουμε σημαντικό ρόλο και κατά το παρελθόν ε, πολλοί έλεγαν ότι οι Άπωνες ε, είναι ιδιαίτερα εθνικιστές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ψάχνει κανείς συγκρίσεις, εγώ να σας πω το εξής. Εγώ ε, ήμουν εισηγητής για τις εταιρικέ σχέσεις στην, στον ελληνικό. μιλάμε για... μια περιοχή ας πούμε, που έχει 1.300 κατοίκους ε, που σημαίνει ότι είναι κατά ένα εκατομμύριο φορές μικρότερο αυτό το νησί, η περιοχή αυτή, από την Κίνα. Απλά το λέω έτσι για να έχετε και μια εικόνα της τάξης μεγέθους, τι ακριβώς πράγμα μιλάμε. Τώρα να απευθυνθώ στην κυρία Γκόμες. Εμείς σίγουρα δεν θέλαμε να ιεραρχήσουμε το πρόβλημα της ασφάλειας ε, ανάλογα με την ε, σημασία του δηλαδή με την έννοια ότι η λάθρομετανάστευση έχει την, ε, βρίσκεται στην ίδια βάση όπως η τρομοκρατία. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα πολιτικής φύσης πρόβλημα και δεν αφορά εμάς. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για να ε, δούμε ή να ισχυριστούμε κατά πόσο η λαθρομετανάστευση ε, δημιουργεί πρόβλημα στην ασφάλεια. Εμείς δεν ζητάμε ένα ε, οχυρό Ευρώπη, αλλά ούτε ζητάμε βέβαια και μια επιθετική και μιλιταριστική πολιτική. Εμείς μιλάμε εδώ για την προληπτική άμυνα ως μια εγγενή αξία, ευρωπαϊκή αξία. Αυτό το περίφημο forward presence, ένα είδος εμπροστοφυλακής αν θέλετε, ε, είναι καθοριστική σημασίας στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Λαντσμπέργκης, μία σύντομη παρατήρηση. Θα ήθελα να ζητήσω μία διευκρίνηση, ε, αλλά δεν, εγώ ζήτησα μία διευκρίνηση, αλλά δεν είπατε τίποτα. Μιλήσατε για υπηρετική ολοκλήρωση. Με ποια έννοια. Μέχρι το 1992... υποτίθεται ότι ήταν αυτή η ολοκλήρωση και μετά ε, ήταν υπερπόντια ολοκλήρωση. Γιατί η πυρωτική μέχρι το 92. Και μετά τι έγινε. Επέκταση μέσα έξω από την Ευρωπαϊκή Ήπερο. Και γιατί μιλάτε για διεύρυνση και όχι, για επέκταση και όχι διεύρυνση. Μήπως έχετε κατά νου ε, κάποιες ε, ειδικές θέσεις σχετικά με τα υπερπόντια εδάφη. Και κατόπιν, όσον αφορά τις ε, στρατιωτικές ε, εγκαταστάσεις της ε, Ρωσίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα γιατί νομίζω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Μιλήσατε για τις προτάσεις που χρησιμοποιήσαμε, για τις λέξεις υπηρωτική ολοκλήρωση», «ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Υπήρου». Εννοούσαμε τη δημιουργία αυτού του οικοδομήματος, καταρχάς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιήσαμε αυτές τις λέξεις για να κάνουμε μια επίσημη περιγραφή της διαδρομής. Εγώ προσωπικώς θα έλεγα ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της λέξης διεύρυνσης και της λέξης ολοκλήρωσης. Η διεύρυνση είναι μια μορφή ολοκλήρωσης ε, ώστε να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη μορφή που έχει σήμερα. Ούτε πιστεύω ότι υπάρχει και μεγάλη διαφορά μεταξύ της επέκτασης και της διεύρυνσης. Το ίδιο πράγμα είναι επέκταση και διεύρυνση κατά την άποψή μου. Ουσιαστικά επεκτείνεται κανείς και κερδίζει άλλους ανθρώπους, άλλες χώρες, άλλα γεωπολιτικά συστήματα επί εθελουσία βάση. Μιλούμε για εθελοντική επέκταση διότι θεωρεί ο κόσμος ότι είναι καλό να μπει κανείς, να μπει ο λαός, να μπει η χώρα η εκάστοτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το επιθυμούν. Εξού και ήδη η προσχώρηση, η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρωμανίας. Δεν ε, είναι όμως μόνο εθελούσια η βάση Δηλαδή δεν είναι και καταναγκαστική, δεν είναι απαραίτητα καταναγκαστική, αλλά είναι μεν εθελοντική, εθελούσια, αλλά υπάρχει και μια δυναμική που σε εξαναγκάζει. γιατί θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να έχει κανείς αυτή τη θέση στο ε, ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Τώρα, ως προς τη Ρωσία, γνωρίζουμε πολύ καλά τι επιδιώκει στο Κάφκασο, στην Κεντρική Ασία και γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλει με αυτή την καινούργια στρατηγική της για τον αρκτικό κύκλο. Και κατανοούμε ότι είναι μεγάλη πρόκληση, αν δεν είναι και απειλή οι βλέψεις όλες αυτές της Ρωσίας. Μπορεί να είναι πρόκληση και απειλή στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Με τις αλλαγές του κλίματος μπορεί να επηρεαστεί ο αρκτικός κύκλος και μάλιστα η υποθαλάσσια περιοχή του αρκτικού κύκλου και ίσως ανοίξουν καινούριες θαλάσσιες διελεύσεις, καινούργια θαλάσσια περάσματα, τα οποία θα καταστήσουν τη Ρωσία πολύ πιο δραστήριο παίκτη στην περιοχή, μια περιοχή στην οποία έχουν συμφέροντα πολλές ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά, και σχετίζεται όλο αυτό με την βόρεια διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής μας. Το γνωρίζουμε, δεν θέλαμε καθόλου να το παραγνωρίσουμε, ούτε να το παραμελήσουμε. Το αφήσαμε λίγο κατά μέρος λόγω έλλειψης χρόνου στην απογευματινή αυτή συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τη δουλειά που κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Μιλούμε για τη δημοκρατική εξέταση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ασφάλεια και την άμυνα. Αυτό είναι το καθήκον το οποίο ασκούμε από κοινού με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, έχουμε διεξάγει δημόσιες συζητήσεις, οι συνεδριάσεις μας είναι δημόσιες και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις εκ του σύνεγγης με το Συμβούλιο. Ε, ο κύριος Μάθιουσον, έχουμε πολύ καλές επαφές με το ΝΑΤΟ αλλά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και νομίζω ότι έχουμε λειτουργήσει σωστά ε, υιοθετώντας την συνολική προσέγγιση των ευρωπαϊκών θεμάτων καταφέραμε να αποκτήσουμε ενημέρωση σε βάθος και με τα ταξίδια μας και με τις αποστολές μας και με τις συζητήσεις, τις ακροάσεις εδώ ε, μετά από πρόσκληση των διαφορών ειδικών και εμπειρογνωμόνων. Αποκτήσαμε στοιχεία και για μυστικές διαδρομές και μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συστάσεις και προσπαθήσαμε κιόλας να εκδώσουμε συστάσεις πριν αποφασιστεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιαδήποτε δράση ή αποστολή στο διεθνές στερέωμα. Και είναι κάτι το οποίο πετύχαμε. Επίσης ασκήσαμε δημοσιονομικό έλεγχο και αυτό είναι ε, ένα από τα λιγότερο γνωστά σκέλη της δουλειάς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξέρετε, γιατί Τέτοιου είδου δράσει και αποστολέ έχουν ήδη ενταχθεί στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί ασκούμε τακτικό έλεγχο και προσπαθούμε να δούμε, να βλέπουμε, να εξετάζουμε τι γίνεται ακριβώ με τα χρήματα των Ευρωπαίων και των προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δουλέψαμε πάνω στις δομές διοίκησης, δουλέψαμε πάνω στον εξοπλισμό, εκπονούμε ιδέες για την ασφάλεια των προσώπων, των ατόμων που εμπλέκονται στις ε, διεθνείς ε, επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συμμετάσχουμε ε, στην καλλιέργεια μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας ασφάλειας και άμυνας Αυτά κάναμε και αυτά είναι αυτά που κληροδοτούμε το επόμενο κοινοβούλιο. Τα μέλη μετά τις εκλογές θα πρέπει να πάρουν τη σκητάλη και να συνεχίσουν αυτό το έργο. Θα ήθελα τώρα να σας καλέσω έξω από την αίθουσα στο χώρο όπου θα πιούμε ένα απεριτίφ και θα έχουμε την ευκαιρία να